Αρχίζουμε τη συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι, λέει ο πρόεδρος. So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας συνάντηση καλωσόρισαν και τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και της Επιτροπής Αναδείξεως και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πάμε τώρα στο πρώτο μας ε, θέμα. Θα πρέπει δηλαδή να εγκρίνουμε τη δημιουργία διάταξη, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις από πλευρά σας, όχι από ό,τι φαίνεται, οπότε εγκρίνεται άνευ μεταβολών. Δεύτερο θέμα είναι οι συνήθειες εγκοινώσεις του Πρόεδρου. Δεν έχω τίποτα εγώ, εκτός από ε, αυτή την κοινή συνεδρίαση ότι θα μεταδοθεί από το ίντερνετ ως συνήθως και υπάρχει και επιτελείο για την τηλεοπτική ε, μετάδοση και έχουμε διερμηνία ε, σε 20 γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμα παριθμών 3 είναι τιμή μου να προεδρεύω κι εγώ αλλά και ο συνάδελφος ο Τωμά και η Μαρία Αρένα τρόπης ε, ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, αντίστοιχα και έχουμε τώρα τον, ε, την εκπρόσωπο του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάροφ. Επίσης έχουμε συνεννόηση και με την αντιπροσωπεία σχέσεων με την Κίνα και επίσης Καλώ όρισε ο κύριο Μπιτικόφερ από αυτήν την αντιπροσωπεία. Δεν μπορούσε να είναι το επομένω ο βραδευτή, αλλά καλώ όρισε η κόρη αυτού. Ε, κυρία Ιλάν, καλώ ορίσατε. Κυρία Ιλάμ, αυτή τη βδομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο έχετε έλθει για να δεχθείτε για λογαριασμό του πατέρα σας αυτό το βραβείο. Είναι δύσκολο, ξέρουμε. Ε, ε, για εσά να μην στεδόχω στον πατέρα σα, για όλα αυτά που έχει κάνει, για αυτού του αγώνε που έχει δώσει με θάρρος ε, το οποίο και εσείς έχετε επιδείξει και όπως ξέρετε ε, απονέμουμε αυτό το βραδύ την ελευθερία της σκέψης από το 1988 και αυτό είναι η απτή απόδειξη του ότι έχουμε δεσμευτεί ε, προς την κατεύθυνση τη πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οπότε αμείβουμε κάποιους αξιοθαύμαστους ε, φορείς ή φυσικά πρόσωπα που δίνουν αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη διότι ακριβώς έχει νόημα αυτός ο αγώνας στο σημερινό κόσμο. Όπως ξέρουμε συνταράσσεται όλη η δρόγιος φέτος από α, διαμαρτυρίες, ε, πολλές φορές και δικαιοσυνη διοτι ακριβως εχει νοημα αυτος ο αγωνας στο σημερινο κοσμο οπως ξερουμε συνταρασσεται όλοι οι δρογιος φετος απο α διαμαρτυριες πολλες φορες και βλέπουμε τι γίνεται στο Χονγκ Κόνγκ, στο Αλγέρια, στο Σαντιάγο Χιλής ε, και σε άλλους τόπους της υδρογείου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο έχουν την ελληνική μας. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι έχουμε τόσα κινήματα τα οποία κάθε μέρα διεκδικούν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Αυτό το έκανε και ο θαραλέος πατέρας σας, ο καθηγητής τότε και ανεγνωρισμένος καθηγητής οικονομικών, να ζωή του στην ε, μειονότητα των Ουιγκούρ στην Κίνα και στα δικαιώματά τους πάνω από δύο δεκαετίες και παλεύει για την αμοιβία κατανόηση Ουιγούρων και Κινέζων. Έχει δημοσιεύσει αναλύσει όσον αφορά τα θέματα κοινωνικά, ε, ε, πολιτικά, οικονομικά, πολιτικά και θρησκευτικά των Ουιγούρων. Το 2006 δε έστησε αυτό το website για την κινέζικη γλώσσα και αυτό ήταν μια πλατφόρμα για ανταλλαγές μεταξύ των Κινέζων, των Χάν και των Ουιγούρων και το κλείσανε και, θεωρήθηκε ότι είναι ηθικός αυτούργος για κάποιες δίες ε, επιθέσεις από ακτιβιστές Ουιγούρους το 2014 καταδικάστηκε σε ισόβια μετά από μια άδικη, εικονική δίκη που κράτησε δύο μέρες. Ε, παραμένει όμως μετριοπαθής και παραμένει υπέρ της συνεννόησης παρά τα όσα έχει τραβήξει. Και με το βραβείο αυτό θέλουμε ακριβώς να ελκύσουμε την προσοχή στα όσα περνά η μειονότητα των ε, Ουιγούρων στην ε, Κίνα. Και τώρα έχει την σκετάλη ο πρόεδρος ε, Τομπέ για λογαριασμό της Επιτροπής Ανάπτυξης από το 2017, συνάδελφοι. Το 2017 λέμε ότι η Κίνα έχει φτιάξει αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, κράτησης. Οι αρχές στην αρχή αρνιόντουσαν την ύπαρξή τους και τα ονόμαζαν ε, κέντρα, κατασκηνώσεις για εκπαίδευση και ε, επανεκπαίδευση και παιδί. Αυτά τα ε, στρατόπεδα είναι απάνθρωπα, είναι απαράδεκτα και εκεί έχουν φυλακίσει, εκεί κρατούνται ένα με δύο εκατομμύρια Ουγγόρων και άλλων μειονοτήτων μουσουλμάνων, οι οποίοι ε, γι' αυτόν τον τρόπο περνούν ε, από κάποιο είδους προσιλητισμό και θέλουν να τους ξεριζώσουν τα πιστεύω τους και η Κίνα τους θεωρεί εξτρεμιστές. Αυτού του είδους τις ε, κρατήσεις, φυλακίσεις, ε, η Κίνα τις θεωρεί ως επιτυχή μέτρα πρόληψης. Όλη αυτή η ιστορία είναι ανατριχιαστική. Το Κοινοβούλιο κατήγγειλε αυτές τις μαζικές καταπατήσεις των δικαιωμάτων των Ουιγούρων. Τρία ψηφίσματα έχουμε εγκρίνει, το 16, το 18 και το 19. Και η σχετική πολιτική της Κίνας επικρίθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στην Τρίτη Επιτροπή του ΟΗΕ το 2019. Παρόλα αυτά, κάποιες χώρες και μουσουλμανικές προέβησαν σε κοινέ διακηρύξεις και δηλώσει υπέρ της Κίνας. Στο πιο πρόσφατο ψήφισμα του 18 η Τετάρτου του 19, το Κοινοβούλιο απίθυνε έκκληση στην κυβέρνηση τη Κίνα άμεσα να απελευθερώσει του Σουηγούρους και τον Ιλαμτότη, τον Τασπολά Ταχύπ, τον Ραχίλ Ενταβούτ και τον Έλλη Μαμούτ και άλλου ε, ηγέτε, κάποιου οι οποίοι είχαν διωχθεί για τι θρησκευτικέ του πεπιθήσει. Όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν κατηγορίε ποινικών δικαστηρίων ή ήδη έχουν φυλακιστεί επειδή άρχισαν το δικαίωμά του ή στην ελεύθερη έκφραση. Και στο ίδιο ψήφισμα το Κοινοβούλιο κατηγορηματικά είχε διατυπώσει την απογοήτευση διότι στον 37ο γύρο 37η δηλαδή, συνάντηση κορυφη Ευρώπη Κίνα. Ε, δεν υπήρξαν αποτελέσματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό καλέσαμε το Συμβούλιο να μελετήσει στοχευμένες κυρώσεις κατά των ε, υπαλλήλων, κατά των Κινέζων αρμοδίων που έλαβαν αυτά τα μέτρα για την αυτόν περιοχή των Ιγούρων. Και σα υπενθυμίζω ότι είναι ο τρίτο Κινέζο ο κύριο τότε ο οποίο ε, αναδέχεται αυτό το γραφείο. Το 1978 είχαμε τον Σέγγ και είχαμε πει ότι πρόκειται τον πέμπτο εξυγχρονισμό και την Κινέζικη Δημοκρατία. Οπότε είχε πάρει αυτό το βραβείο ένα χρόνο πριν. Ε, αποφυλακιστεί και εξοριστεί στην Κίνα το 2008 Χουτζία που ήταν ε, ένας ακτιβιστής ο οποίος ε, τρία χρόνια πριν είχε αποφυλακιστεί και έχουμε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατο που είχε σχολιάσει τον τότε ο κύριος Χουτζία και είχε πει ότι αυτό μόνο που θέλει ο κύριος τότε είναι ισότητα, αξιοπρέπεια και ειρηνική συνύπαρξη για τον λαό του. Και αν η κοινωνική κυβέρνηση τον θεωρεί ότι είναι αποσχιστής, ε, είναι σαν να λέω ότι όλοι οι Γούροι είναι τρομοκράτες. Εμείς, ε, κυρία μου, θα συνεχίσουμε να υπερσπιζόμαστε τον πατέρα σα και να διεκδικούμε την ε, άμεση αποφυλακή σου. Και τώρα, ισχυτάλη στην κυρία Ερενά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα γαλλικά. κυρία ελάμ όπως είπε ο συνάδελφος Τομπέ, μπορείτε να υπολογίζετε σε εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να καταλάβετε ότι εμείς κάθε φορά που μπορούμε να το κάνουμε θα ζητούμε να, αφήνετε, να αφαιθεί ελεύθερος ο πατέρας Στο μέλλον σε όλες μας τις σχέσεις με την Κίνα. Απονέμουμε αυτό το βραβείο φάρο για εκείνους που ενσαρκώνουν την αντίσταση και την ελευθερία ο πατέρας σας είναι άνθρωπος του διαλόγου και του ανοιχτού πνεύματος. Γνωρίζουμε ότι το βραβείο Ζαχάροφ ε, δημοσιοποιεί ε, ε, τα αιτήματα, προβάλλει τους βραβευθέντες και εκνευρίζει τις κυβερνήσεις, οι οποίες κατηγορούν για επέμβαση στα εσωτερικά τους. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι κριτικές. Το Κοινοβούλιο οφείλει να παραμείνει ε, σε επιστράτευση για όλους τους κατόχους του βραβείου Ζαχάροφ που παραμένουν στη φυλακή και να ε, πλησιώνει εκείνους που συνεχίζουν αυτή την ευγενή ε, μάχη που δίνουν. Το 2019 είχαμε καλά νέα, διότι αφέθηκαν ελεύθεροι δύο βραβευθέντες. Το 2007 ο Σαλίος Μάρν που επανειλημμένα τον είχε φυλακίσει το δικτατορικό καθεστώς του Σουδάν αρχές του έτους αφέθηκε ελεύθερος μετά τις ε, πολιτικές ε, ε, αναταραχές στη χώρα. ήρθε ελεύθερος στην Επιτροπή μας, υπό Επιτροπή Ντρουά, τον περασμένο Οκτώβριο. Μας έκανε αυτή τη τιμή. Πριν από ένα μήνα, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, υποδεχτήκαμε στο Στρασβούργο, εδώ στην αίθουσα, τον Ουκρανό κινηματογραφιστή ε, Όλεκ Σέντσοφ, που τιμήθηκε πέρσι με το βραβείο. Ήταν ενώπιόν μας επιτέλους ελεύθερος και είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψη για την κατάσταση στη χώρα του. Δυστυχώς την περασμένη εβδομάδα μάθαμε ότι ο Ραΐφ Μπαντάουι ε, που πήρε το βραβείο το 2015 άρχισε απεργία πείνας γιατί τον μετέφεραν ε, στην απομόνωση στη φυλακή που βρίσκεται μαζί με τον συνήγορό του. Καλούμε τις αρχές του Ριάντ να σταματήσουν αυτή την παρενόχληση και να τον αφήσουν αμέσω ελεύθερο και τον ίδιο και τον συνήγορό του. Ε, θέλω να θυμίσω την Αστρίν Σατούντε ε, που το 2012 ήταν εκ των βραφευθέντων ε, και πάλι τη συνέλαβαν στο Ιράν και την καταδίκασαν σε 38 έτη κάθερξη. Αυτό είναι ακατανόητο και ε, απερίφραστα το καταδικάζουμε. Ραζάμ Σατουνέ από την Αραβική Άνοιξη νεαρή δικηγόρος από τη Συρία. 7 χρόνια δεν έχουμε νέα της σχεδόν καθόλου. Θα πρέπει λοιπόν να τιμούμε αυτές τις ιδιαίτερες προσωπικότητες. Συμμεριζόμαστε κοινέ ανθρωπιστικές αξίες και είναι στον πυρήνα και την καρδιά της Ευρώπης. Θα πρέπει να είμαστε στο ύψος αυτών των αγώνων, δηλαδή συνεπείς στις πολιτικές μας. Και μιλώ εδώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στην Επιτροπή αυτή. Έχουμε και την Επιτροπή Εξωτερικών και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Όλες όμως οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μας θα πρέπει να ενσωματώσουν στη δράση τους τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην παγκόσμια δράση τους. Παρακαλώ βεβαιωθείτε κυρία μου ότι αυτό το βραβείο Ζαχάροφ θα μας συνδέει μαζί σας και με τους αγώνες του πατέρα σας μέχρι να φεθεί ελεύθερος και ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα να γίνει γεγονός αυτή η ε, απελεύθερωση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μαρία Ρένα. Σε ευχαριστώ το μας τον Μπέ και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με μεγάλη μου τιμή δίνω το λόγο στην κυρία Τσανχέρ Ιλάμ ε, κόρη του καθηγητή Ιλάμ Τότη που ε, βραβεύθηκε με το βραβείο Σαχάρο φέτος το 2019. Καλησπέρα σας. Ε, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ζαχάρ Ιλάμ. Δεν έχω ετοιμάσει ομιλία σήμερα. Θα σας μιλήσω με την ιδιότητα της κόρης ε, του ανθρώπου αυτού και μέλος μιας κοινότητας. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω αφού σας αφηγηθώ κάποιες ιστορίες, Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο που απένιμε το βραβείο ζαχαρο στον πατέρα μου. Ε, δεν μπορούσε να βρίσκεται φυσικά εδώ για να ε, έχει ο ίδιος το βραβείο να πάρει ίδιο το βραβείο στα χέρια του. Ε, ε, θα ήταν πραγματικά ε, το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά γι' αυτό μετέδινα εγώ. Αυτό που εύχομαι πάνω απ' όλα, ένα τέτοιο βραβείο, να μην είχε λόγο ύπαρξης στον κόσμο μας σήμερα. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα είχαμε και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω κάποτε να μην υπάρχει κανείς που θα πρέπει να χρειάζεται να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ανακτιβιστεί. Πραγματικά εύχομαι να απελευθερωθεί ο πατέρα μου και όλοι οι ακτιβιστέ, όσοι έχουν βεβαιωθεί όχι όπω ο πατέρα μου, ε, να απελευθερωθούν. Τώρα, τι άνθρωπο είναι ο πατέρα μου. Είναι φιλότιμο. Είναι πολύ θαραλέος και με μεγάλη καρδιά. Του συγχωρεί όλους. Προτού συλληφθεί, θυμάμαι μια φορά σε μια από τις συνομιλίες μας στο Skype μου είπε «Κορή, έχω την εντύπωση ότι μπορεί σύντομα να συλληφθώ». Και τότε, αν συμβεί αυτό, μην ε, θα παίξει, μην φοβηθείς, μην μισήσεις την κινέζικη κυβέρνηση. Δεν θέλω να ζεις μες στο μίσος». Και αυτό που υποστηρίζει η κινέζικη κυβέρνηση και όλοι γύρω μου είναι ότι είναι αποσχιστή ο πατέρα μου. Κι όμω αυτό που ζητά είναι να μην υπάρχει βία. Δεν είναι εξτρεμιστή. Θα έλεγε ποτέ ένα εξτρεμιστή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Είναι απλώ κάποιο. Μάλλον είναι κάτι που θα έλεγε. Είναι κάτι τέτοιο αυτό που θα έλεγε ένα ε, προασπιστή τη βία. Δεν νομίζω. Υπήρξαν και άλλε περιπτώσει όπου ο πατέρα μου χρησιμοποίησε ένα όπλο τα λόγια του. Με το λόγο του προσπάθησε να προτείνει λύσεις για προβλήματα. Προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα στην Κίνα και δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Ο πατέρας μου πίστευε και πιστεύει ότι έναν επίλυτο πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκείνος ήθελε να βρει λύσεις. Ήθελε να διευκολύνει την κινέζικη κυβέρνηση γιατί έβλεπε τα προβλήματα και πίστευε ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι μπορεί να λυθούν τα προβλήματα. Ήθελε λοιπόν να βοηθήσει και όχι να δυσκολέψει τα πράγματα. Όμως αντί να γίνουν δεκτές οι λογικές και μετριοπαθείς ε, συμβουλές του, τελικά τον έστειλαν στη φυλακή και τον καταδίκασαν σε ισόβια. Σε μια από τις συνεντεύξεις του, ο πατέρας μου είπε «Γνωρίζω ότι θα μπω φυλακή. Το ξέρω. Ίσως να καταδικαστώ σε δεκαετή Κάθερξη ίσως σε 20 χρόνια. Αλλά η κινέζικη κυβέρνηση κάπου θα σταματήσει, δεν θα κάνει και πολύ, κάτι πολύ χειρότερο. Και όταν βγω έξω, θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο. Θα συνεχίσω να βοηθάω του ανθρώπου τη κοινότητά μου και του Κινέζου. Αυτά έλεγε ο πατέρα μου. Τέτοιου είδου άνθρωπο είναι. Και είμαι 100% πεπισμένη ότι αν υπήρχε μηχανή του χρόνου και ο πατέρα μου μπορούσε να πάει μια πενταετία πίσω όταν ε, συνελήφθη πρώτη φορά, πριν από τη σύλληψή του ακριβώς θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Θα συνέχιζε να αγωνίζεται για την κοινότητά του, για το λαό μας. Ακόμη και αν ήξερε ότι θα καταλήξει τελικά στη φυλακή και μπορεί και να ε, πεινάει μέχρι θανάτου ε, στο σκοτεινό και υγρό κελί του δεν με εκπλήσει, ούτε θα μου έκανε εντύπωση κάτι τέτοιο, γιατί τέτοιο άνθρωπος είναι. Τα τελευταία πέντε χρόνια προσπαθώ με κάθε τρόπο να προβάλλω την περίπτωση του πατέρα μου, την υπόθεσή του και εδώ και ένα χρόνο έχω συνεργαστεί με πολλού ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολλέ οι φορέ που είπα θα τα παρατήσω. Δεν αντέχω να πάρω μέρο σε άλλη συνεδρίαση και σε συνάντηση. Δεν μπορώ να περνάω όλη μου τη ζωή σε αυτό. Το έχω πει ξανά και ξανά, όμως να είμαι πέντε χρόνια μετά, εδώ μπροστά σας, παρόλο που ξέρω ότι η συνεδρίαση αυτή, η συνάντηση αυτή και το βραβείο αυτό μπορεί πραγματικά να προκαλέσει την ε, οργή της κινέζικης κυβέρνησης. Αλλά οφείλω να το κάνω. Δεν μπορώ να παρατηθώ, δεν μπορώ να μείνω αδρανής. Διότι εάν το κάνω αυτό δεν θα μπορώ να ξαναντικρίσω τον πατέρα μου. Θέλω να είναι υπερήφανο για μένα και θέλω να είναι υπερήφανο για τον εαυτό του που ε, με μεγάλωσε, με ανέθρεψε και με έφτιαξε ε, όπω είμαι σήμερα. Ο καθένα σε αυτή την αίθουσα αυτό που μπορεί να κάνει είναι να συμμετέχει. Παρακαλώ βοηθήστε τον πατέρα μου. Βοηθήστε τους εκατοντάδες ε, εκατομμύρια, τους δεκάδες εκατομμύρια Ουιγούρους που είναι αθώοι και είναι κλειδωμένοι σε ένα στρατόπεδο, σε μια φυλακή, βοηθήστε τους. Υποστηρίξτε τον αγώνα μας. Διότι ελπίζω και πιστεύω ότι κάτι θετικό θα γίνει μετά από αυτή τη συνάντηση, από αυτή την εκδήλωση σήμερα. Ελπίζω και το εύχομαι ολόψυχα, ε, ας αγωνιστούμε όλοι μαζί. Δεν είναι για έναν φυλακισμένο, δεν είναι για μια κοινότητα, δεν είναι για έναν λαό. Είναι ανθρωπιστικό το θέμα, αφορά τους πάντες. Αφού αυτό συνέβη σε μένα και στη δική μου οικογένεια, μπορεί να συμβεί στην οποιαδήποτε οικογένεια, στον καθέναν σε αυτόν τον πλανήτη. Και είναι στιγμή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ε, κύριε Ελχάμ. Ήταν πολύ προσωπικά τα λόγια σας και πολύ συγκινητικά ταυτόχρονα. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, σε κάποιους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το ζήτησαν και αρχίζω από τον κύριο Πίτσι Κόφερ που είναι ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κίνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ilham. Σας ευχαριστώ κυρία Ilham για τα συγκινητικά σας λόγια και σας ευχαριστώ που ήρθατε να παραλάβετε το βραβείο εξ του πατρός σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει για να τιμήσει τις υπηρεσίες του πατέρα σας στην ε, συμφιλίωση, την ελευθερία του λόγου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μαρτυρία σας για τον αγώνα που δίνει ο ίδιος. Δηλαδή, ακόμα και όταν έρχεται αντιμέτωπος με κατασταλτικές πολιτικές από πλευράς ε, του Κινέζικου κόμματος κράτους, συνεχίζει να ζητάει τη συμφιλίωση Πραγματικά θέλουμε να το τιμήσουμε γιατί με το παράδειγμά τους αισθανόμαστε πολύ ταπεινοί μπροστά του. Ταυτόχρονα απονέμουμε το βραβείο Ζαχάρο φέτος ε, στον πατέρα σας. Και αυτό ρίχνει άπλετο φως στην κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα. Στην εθνότητα αυτή στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του πατέρα σα. σας. Και τώρα εφίσταται καταστολή αυτή η, κοινότητα, η εθνότητα με διάφορους τρόπους. Και υποφέρουν από το χειρότερο αστυνομικό κράτος που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη. Και θα θέλαμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τη συμπόνια μας προς τους ανθρώπους αυτούς που διώκονται γιατί ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη εθνότητα ή σε κάποια θρησκευτική κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν πολύ στεναρά ετώνιζε και υπογράμμιζε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μας τους Ευρωβουλευτές η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στην ίδια την καρδιά της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι στα γονίδια μας τα πολιτικά. Συνεχώς λοιπόν και σε τακτά χρονικά διαστήματα ασχολούμαστε με τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή του πατέρα σας. Σε περιπτώσεις άλλων ουγγούρων ή άλλων μουσουλμάνων στην Κίνα και στο Σιντζάν και πανταχού της γης που υφίστανται αυτή την καταπίεση. Στόχος μας δεν είναι μόνο η αύξηση της συνειδητοποίησης, αλλά και η ανάληψη δράσης για να μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτούς τους δύσκολους αγώνες που δίνουν. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ένα παγκόσμιο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων για λόγους παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν υπάρχει καν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω είναι πολύ θετική εξέλιξη ότι ο νέος ύπατος εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο νέος ας πούμε, Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μπορέλ, μετά το τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων είπε ότι και τα μέλη του Συμβουλίου τώρα προχωρούν προς μια τέτοια σκέψη να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων παγκοσμίω για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε, χρειάζεται να συμφωνήσουν και οι δύο συνομοθέτες, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, για να γίνει η νομοθεσία αυτό. Πάντως, ευελπιστούμε ότι μπορεί να ευοδοθεί αυτή η προσπάθειά μας ενδεχομένως του χρόνου. Και αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε ακόμα πιο στεναροί στη δράση μας και στην προσπάθειά μας και να υποστηρίζουμε τους αγώνες αυτούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου και αν συμβαίνουν. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για όσα κάνετε, για την πίστη που εκφράζετε στις αρχές που όλοι ε, συμμεριζόμαστε και Εύχομαι η οικογένειά σας να ξαναδεί τον πατέρα σας σύντομα ελεύθερο και υγιή, ελπίζω. Ευχαριστώ. Thank you, Reinhard ε, Κύριε Μπουτικόφερ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε τον λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Τρία λεπτά, έκαστος Γκάλερ, για το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα συγκινητικά μας είπατε παρουσιάζοντας τον αγώνα του πατέρα σας, τη διαδρομή του ε, όλη ε, του την ε, ζωή. Πρόκειται για κάποιον που έκανε αγώνες κομμένους και ραμμένους για αυτό το βραβείο. Βεβαίως, παρά τις απειλές που έχει δεχθεί, βροντοφωνάζει την γνώμη του διαδίδει αυτόν τον ε, θεμητό αγώνα και στην Κίνα και σε όλο τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι όπως και άλλοι που έχουν να κερδίσει αυτό το βραβείο, ήταν για το βραβείο, σίγουρα και το αξίζει. Εμείς από αυτή τη θέση στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Όχι βέβαια μόνο με την απονομή του γραφείου, αλλά και συζητώντας για το τι γίνεται με τους ε, Ουιγούρους. Έχουμε φτιάξει αυτά τα ψηφίσματα, έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε ξεκάθαρα τοποθετήσει, έχουμε ξεκάθαρα απαιτήσει μάλλον ε, από τους Κινέζους ότι αυτά τα οποία λένε δεν στέγουν δηλαδή ότι πρόκειται για εθελούσια συμμετοχή αυτών που βρίσκονται σε αυτά τα στρατόπεδα για να εκπαιδευτούν και ότι θα έπρεπε, του έχουμε πει, να έχουν διαφάνεια, να, έχουν, να αφήσουν δημοσιογράφου, να αφήσουν τον ΟΗΕ και οργανώσει ε, δικαιωμάτων εκεί να επισκεφτούν και να δουν για να ζυγίσουν πώ έχει αυτή η κατάσταση με αυτού που είναι εκεί κλεισμένοι. Αλλά βέβαια αυτοί άλλα πρεσβεύουν. Πρόκειται για εκατομμύρια, για κάνω οι οποίοι είναι υποπεριορισμό. Φυσικά και πρέπει τη θέλησή του. Όμως, με διαφάνεια και με ανοιχτό πνεύμα θα έπρεπε να διερευνηθεί η τύχη αυτών των ανθρώπων. Όσον αφορά αυτά τα στρατόπεδα, έχουμε παραγωγή αγαθών που εξάγονται, εξάγονται σε διάφορες χώρες. Ε, αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε. Καμία κινέζικη εταιρεία εξαγωγών τέτοιων προϊόντων που είναι από το καταναλωτική εργασία να μην βρίσκει διέξοδο για τα προϊόντα της στην Ευρώπη ή αλλού. Σε αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί. Και θέλω να σας ρωτήσω. Ξέρετε τίποτα σχετικά. Έχετε κάποια στοιχεία για τέτοιες πρακτικές. Εκτό από τον ε, πατέρα σας ε, μπορούν οι ε, δικηγόροι να βοηθήσουν τον κόσμο σε αυτά τα στρατόπεδα. Ναι, ξέρουμε ότι ο πατέρας δεν βρίσκεται σε αυτά τα ε, αναμορφωτήρια, στα πούμε έτσι, σε μια κανονική φυλακή, αλλά λέμε για εκείνα τα στρατόπεδα. Οπότε, αν μπορούσατε, πέστε μας κάποια παραπάνω στοιχεία, αν έχετε κάτι ακούσει. Θα ήταν δυνατόν να υπάρχει κάποια ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στην Κίνα, κάπως να υπάρχει κάποια επικοινωνία και μεταξύ αυτών των ατόμων. Ευχαριστώ με... έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ε, βέβαια, πρώτα απ' όλα και συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το σύστημα, σε αυτά τα αναμορφωτήρια. Και βέβαια με τίποτα δεν με πείθει ότι ο χαρακτήρας τους είναι εκπαιδευτικός. Ούτε έχει καμία σχέση με εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση, με σχολείο. Αν ήταν έτσι θα μπορούσε ο κόσμος να πάει σπίτι του αν ήθελε. Και να πει ένα πρωί που δεν αισθάνομαι καλά, σήμερα θα πουσιάσω από το σχολείο. Αλλά ο κόσμος που είναι εκεί πολλές φορές είναι πάνω από 70 ή κάτω από 20. Πολλοί από αυτούς είναι καθηγητές πανεπιστημίων. Κάποιοι έχουν αξιόλογες εργασίες όπως είναι γιατροί, ε, τεχνικοί πληροφορικής, ε, ε, προπονητές ε, δεν, δεν έχουν ανάγκη από επανεκπαίδευση. Μετεκπαίδευση τέλος πάντων. Και ε, θα μπορούσε να ελκύσει την προσοχή άλλων χωρών η Κίνα. Για να δούμε τι γίνεται στην Κίνα, τι γίνεται με τους Ουιγούρους, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος τι γίνεται εκεί. Πρόκειται για την ίδια χώρα, αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος εκεί, οι Κινέζοι, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε κανονικά ΜΜΕ, μια που υπάρχει λογοκρισία full. Μιλήσατε για τις κυρώσεις προς ε, τις εταιρείε εκείνες και συμφωνώ μαζί σας. Όχι, όχι, δεν λέω να επιβληθεί γενικά ε, μέτρο ε, προς την Κίνα γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαία χώρα, έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ σημαντικό η κάθε χώρα να μπορεί να συνεργαστεί και να υπάρχει κέρδος οικονομικό και ωφέλεια για τους ε, πολίτες. Αλλά παντού οι χώρες να μην εκβιάζονται από την υπόθεση αυτή του οικονομικού ωφέλους. Αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτές τις εταιρείες που ωφελούνται από αυτά τα στρατόπεδα. Και για την άλλη ερώτησή σας, από ό,τι έχω μάθει, ήταν στην απομόνωση ο πατέρας μου. Ήταν στην πρώτη φυλακή του Ρούμτσι. Τελευταία φορά τον επισκεφτήκαμε το 17. Σύμφωνα με το συνέγμα της χώρας, δικαιούνται κάθε μήνα επίσκεψη φυλακισμένη. Για τον πατέρα μου όμως αυτό ήταν τρίμηνο στην αρχή. Και από το 17 άπαξ και ε, ξέφυγε η κατάσταση με τα στρατόπεδα, δεν έγινε καμία επίσκεψη, οπότε δεν ξέρω που είναι. Αν ακόμα είναι σε φυλακή ή αν έχει μεταχθεί σε κάποιο τέτοιο στρατόπεδο, σε άλλο είδους κέντρο κράτησης, ούτε αν είναι ζωντανός δεν ξέρω. Οπότε θα ήταν υπέροχο εάν οι ηγέτες διαφόρων χωρών μπορούσαν να πιέσουν την Κίνα. Βεβαίω να τον αποφυλακίσει, αλλά τουλάχιστον να μας πούν σε εμά στην οικογένειά του πού είναι, τι κάνει, αν ζει. Δεν είναι τόσο δύσκολο για την κινέζικη κυβέρνηση και σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας οφείλουν να το κάνουν αυτό. Θα πρέπει να επιτρέψουν την επίσκεψη στην οικογένεια. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές η κυρία Σάντους. Ε, παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω πορτογαλικά, όσοι χρειάζεστε βεβαίω μετάφραση. Πάνω απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Ιλάμ για τον αποφασιστικό και τολμηρό τρόπο με τον οποίο από την αρχή προασπίζεστε τον αγώνα του πατέρα σας, ε, τον αγώνα του για ελευθερία και τον αγώνα για απελευθέρωση των Ουιγούρων, ε, για να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί αυτοί είναι οι όροι που αρμόζουν. Ε, είναι πραγματικά ε, κάτι που μας σοκάρει και είναι κάτι που ήταν ε, βάναυσο ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο πατέρα σας και το πώς εσείς χρειάζεται να αγωνιστείτε για την ελευθερία κάποιου την ελευθερία κάποιου που το μόνο που έκανε ήταν να χρησιμοποιήσει το όπλο των λόγων του. Ένα όπλο πολύ επικίνδυνο βεβαίω να χρησιμοποιηθεί σωστά. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ και τον ε, πατέρα σα ε, για το θάρρο του, γιατί ήταν πάντοτε ένα άνθρωπο διαλόγου με ανοιχτό πνεύμα που πολέμησε για τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ελευθερία. Ένα άνθρωπο που ακόμα σήμερα, ε, ό,τι σε ό,τι συνθήκε και αν ζει, είμαστε βέβαιοι ότι συνεχίζει με το ίδιο πνεύμα να κινείται με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια ενέργεια για να προσπιστεί και να υπερασπιστεί το λαό του. Ε, ό,τι συμβαίνει στην Ξινγιάνγκ είναι πραγματικά απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για στρατόπεδα επανεκπαίδευση, αναμορφωτήρια. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την ε, πολιτιστική γενοκτονία των οιγούρων. Αυτό που έχει επιβληθεί στο λαό των οιγούρων και που πραγματικά συνεχίζει να επιβάλλεται και στο λαό του Θιβέτ παρά τη λιγότερη προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό έχει γίνει ένα μοτίβο, έχει γίνει ένα μοντέλο που ακολουθεί συστηματικά η Κίνα και το καθεστώς της. Ένας άνθρωπος που αντιστάθηκε σε αυτό το πρόγραμμα καταστολής του Θιβέτ ε, έχει την ίδια μοίρα με τον άνθρωπο που ύψωσε το ανάστημά του στο καθεστώς ε, καταστολής του Ε, Πραγματικά δεν μας εκπλήσει και ξέρουμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέτρα που συζητούνται και μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτές τις παραβιάσεις, πράγματα που ελπίζουμε να ε, εγκριθούν σύντομα και να υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, αυτό που σημαίνει η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι ότι προβάλλει το κύρος του βραβείου Ζαχάροφ και η μόνη ερώτηση που θέλω εγώ να κάνω είναι τι είδους κυρώσεις μπορείτε να θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσουν για να περιοριστούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ευχαριστούμε, Ιζαμπέλ Σάντου. Θα θέλατε να απαντήσετε απευθεία. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Οχ. Καταρχάς, εγώ πολιτικός δεν είμαι. Δεν ξέρω πώς κυβερνάς μια χώρα. Αλλά η Κίνα είναι μια ισχυρή χώρα. Μπορεί να μην φοβάται μία άλλη χώρα, δύο ή δέκα, αλλά όταν οι υπόλοιπες χώρες συμμετέχουν και σε μια προσπάθεια και είναι ενωμένες και απευθύνουν έκκληση στην Κίνα να τους αφήσει ελεύθερους ανθρώπους αυτούς, σίγουρα θα ακούσει η Κίνα. Ε, υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι, χέφρονες στην ε, κινέζικη κυβέρνηση και ορισμένοι από αυτούς σίγουρα θα ορθώσουν το ανάστημά τους και θα δώσουν μια συμβουλή και θα πούνε «Κοιτάξτε, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος όλος εναντίον μας» και ζητούν να αλλάξουμε τακτική. Για αν δεν το κάνουμε θα υποστούμε μεγάλες κυρώσεις. Και νομίζω ότι η Κίνα θα το πάρει σοβαρά αυτό υπόψη. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερες χώρες. Όχι μόνο η ΕΠΑ, όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά όλες οι χώρες του κόσμου. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι πολίτες. Όλες οι κυβερνήσεις. Αλλιώς η Κίνα θα κάνει ό,τι καπνίζει. Αν ενωθούν όλοι εναντίον της, δεν μπορεί να είναι μοναχικός καβαλάρης. Φιλ Μπένιν και Κιουτσούκ από την ομάδα Ρινιού, 1,5 λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Μπάνιον. Ε, κυρία Ιλχάμ, ο κύριος Κιουτσούκ και εγώ συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια και την εκστρατεία από το 2017. όταν πήρε το φιλελεύθερο παγκόσμιο βραβείο για την ειρήνη ο πατέρας σας. Και τότε είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι φήμες για τα στρατόπεδα αυτά τα αναμορφωτήρια. Και όλο και περισσότερο είχαμε στοιχεία από αυτόπτες μάρτυρες. Ε, συζητήσαμε με ανθρώπους που είχαν δει αυτά τα στρατόπεδα και δημοσιογράφους που πρόσφατα ε, το έφεραν αυτό υπόψη μας. είναι πραγματικά η μοναδική τέτοια έκταση και κλίμακα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω. Γι' αυτό ε, επέμεινα τόσο πολύ με την συγκεκριμένη υποψηφιότητα και θέλησα να περάσει. Η Κινέζικη Πρεσβεία στο Λονδίνο με κάλεσε σε συνεδρίαση για να το συζητήσουμε και μου ζήτησαν να αποσύρω την υποψηφιότητα. Και τους είπα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μα μου είπαν ότι ο άνθρωπος είναι εγκληματία, είναι αποσχιστή, αυτόν υποστηρίζεται. Και θα τον βραβεύσετε και όλα τους ανθρώπου. Αλλά εγώ τους ρώτησα και δεν μου απάντησαν αρνητικά. Ήταν Μήπως θα μπορούσατε να αποκαταστήσετε τα δικαιώματα της οικογένειάς του να τον επισκέπτεται και το συνήγορό του. Κανείς δεν ξέρει αν έχει διψυχία ο άνθρωπος τα τελευταία δύο χρόνια από επισκέψεις. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά να πιέσουμε να γίνει. Γιατί νομίζω ότι εκεί μπορεί να βοηθήσουμε να επιτευχθεί κάποια πρόοδος. Εσείς πώς λέτε να συμπεριφερόμαστε προς τους Κινέζους για να αποκατασταθεί το δικαίωμα επίσκεψης. Και αν φτάσουμε μέχρι εκεί, μπορεί να φτάσουμε και μέχρι την απελευθέρωση. Το έχουμε δει και από άλλους ροβεφέντες. Ο κύριος Κιουτσούκ, ο κύριος Μπάνιεν μίλησε εξ ονόματος της ομάδας μας και χαίρομαι που ακούω ότι σας υποστηρίζουν πολύ το θέμα των, ε, της μειονότητας των Ουγγούρων που ζουν στον Σιντζάκ. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, παρόλο που δεν έχετε νέα από τον πατέρα σας από το 2017. Ούτε εμείς ξέρουμε για τις συνθήκες κράτησης. Χαίρομαι που είστε αισιόδοξοι και επιμένετε. Είναι μοναδικό το παράδειγμα του πατέρα σας και το ακολουθείτε κι εσείς. Νομίζω είναι πολύ σημαντική αυτή η αποκατάσταση των δικαιωμάτων επίσκεψης για μας. Φυσικά θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε και να ζητούμε εμείς μαζί με άλλους να αφαιθεί ελεύθερος. Εσείς πώς βλέπετε τη συνεργασία με την κινέζικη κυβέρνηση. Μετά την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι μπορεί να αλλάξει το βραβείο αυτό κατά τη γνώμη σας. Με ρωτάτε πολύ δύσκολα πράγματα. Δυστυχώς, εγώ δεν εργάζομαι για την κινέζικη κυβέρνηση, ούτε μπορώ να προβλέψω πώς σκέφτονται. Πάντως, εγώ είμαι υπεραισιόδοξη και υπερθετική όπως και ο πατέρας μου και πάντα ελπίζω στο καλύτερο ως έκβαση Και αυτό ήταν για μένα κινητήρια δύναμη μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε πώς έχει η κατάσταση. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Even though my family... Ακόμα και αν η οικογένειά μου ας πούμε αποκτήσει το δικαίωμα να τον επισκεφθεί. Φοβούνται πάρα πολύ να επιστρέψουν στην περιφέρεια εκεί που ζουν οι Ουιγούροι, ακριβώς λόγω των στρατοπέδων συγκέντρωσης γιατί έχουν συλλάβει συγγενείς μου ας πούμε η ε, ξαδέρφη μου που είναι νοσοκόμα ε, συνελήφθη και της επιβλήθη ποινή 10 ετής γιατί είχε στο κινητό της ε, τη φωτογραφία του πατέρα μου. Ο κόσμος φοβάται και η οικογένειά μου φοβάται να επιστρέψει εκεί γιατί φοβούνται ότι θα του συλλάβουν. και ένα συγγενή μου έχει φύγει τώρα στι ΗΠΑ, είναι εκτός Κίνα. Καλό θα ήταν να υπάρχει δυνατότητα για τακτικές επισκέψεις, αλλά μπορεί η οικογένειά μου να επιστρέψει στην περιοχή των Ουιγούρων χωρίς να φοβάται ότι μόλις πατήσει το πόδι της εκεί θα ε, συλληφθεί και θα τις ρίξουν στα ίδια στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ποιο θα του απαλλάξει από αυτό το φόβο. Όλα αυτά συνδέονται τα θέματα. Φυσικά θα ήταν καταπληκτικό εάν ε, επιτραπούν τακτικές επισκέψεις από την οικογένεια. Ο αδελφός μου μόλις έκλεισε τα 13. Ζει στο Πεκίνο και φοβάται να βγει από τη γειτονιά του. Φοβάται να κυκλοφορήσει. 13 χρονό παιδί. που είναι στο άνθος της ηλικία του. Όλοι του οι φίλοι βγαίνουν το καλοκαίρι, το χειμώνα, στις διακοπές. Εκείνος σημαίνει κλεισμένο στο διαμέρισμά μας στο Πεκίνο γιατί είναι κατατρομοκρατημένος, φοβάται ακόμα και να βγει. Πού να γυρίσουμε πίσω στη περιοχή μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Εδώ δεν μπορούμε να βγούμε από τη συνοικία που μένουμε στο Πεκίνο. εδώ και χρόνια δεν έχω μιλήσει με μέλη της οικογένειάς μου γιατί φοβούνται να μου μιλήσουν. Γιατί φοβούνται ότι μόλις μου μιλήσουν θα τους ε, διώξει η κυβέρνηση. Η κινέζικη κυβέρνηση μπορεί να σας υποσχεθεί ότι θα αφήσει τους συγγενείς να επισκέπτονται τον πατέρα μου. Και με μεγάλη χαρά θα την ακούσω αυτή την είδηση. Και μακάρι να έρθει εκείνη η μέρα. Και συγγνώμη, αλλά ξέχασα την ερώτησή σα, κύριε Κιουτσούκ. Μήπω θα μπορούσατε να την επαναλάβετε. Για το βραβείο Ζαχάροφ ρώτησα και πώ ε, ε, θα το εκλάβει αυτό η κινέζικη κυβέρνηση και τι μπορεί να αλλάξει. Ναι, όπως σας είπα και στην αρχή, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και θετική και ελπίζω να έχει θετική επιρροή αυτό το βραβείο για την υπόθεση του πατέρα μου και γενικότερα την κατάσταση των Ουιγούρων. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι θα επιτύχει αυτό το βραβείο. Πάντως είμαι βέβαιη ότι θα, ε, θα συγκεντρώσει την προσοχή, ε, την παγκόσμια στο πρόσωπό του. Και αυτό έχει σημασία. Ότι θα συνειδητοποιήσουν και άλλες χώρες ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βράβευσε τον πατέρα μου ως αναγνώριση του αγώνα των Ουιγούρων και της κατάστασής τους. Και μπορεί και άλλες χώρες να συμπαραταχθούν σε αυτή την προσπάθεια και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ως κίνηση και για άλλες κυβερνήσεις, για άλλους ηγέτες και ελπίζω να βοηθήσει αυτό και την κινέζικη κυβέρνηση να καταλάβει ότι χρειάζεται να παίρνει καλύτερες αποφάσεις. Ελπίζω τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I understand, spoken also for the, on Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μπουτικόφερ κανονικά θα πρέπει να πάρει το λόγο από τους πρασίνους, αλλά ήδη έχει μιλήσει. Από την ID δεν έχουμε κάποιον, οπότε για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, κυρία Φωτίγκα και ο κύριος Τέτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ήλχαμ, που είσαστε εδώ για να μας ε, εκθέσετε τις απόψεις σας. Και ευχαριστούμε που είστε εδώ αποτείοντας φόρο τιμής στον ευγενή πραγματικά και θαραλέο αποφασιστικό πατέρα σας. Είστε και εσείς πραγματικά μία ε, πολύ καλή εκπρόσωπος που μπορεί να εκφράσει τον αγώνα του και να τον προβάλλει για, για εκείνον και το λαό σας. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν υποφέρει και από το κομμουνιστικό σύστημα ε, και καταλαβαίνω γιατί είμαι από την Πολωνία, έχω τα δικά μου βιώματα, τις εμπειρίες της οικογένειάς μου, του λαού μου. Και εμεί ζήσαμε τα ίδια με αυτό το σύστημα και πραγματικά είμαι βεβαία ότι το βραβείο Ζαχάροφ μπορεί λίγο να αλλάξει τη ζωή του πατέρα σας. Και πιστεύω ότι η πίεση που θα ασκήσουμε όλοι μαζί μπορεί να κάνει θαύματα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει γιατικό ρόλο για να αποκαλύπτει αυτό του είδους τις υποθέσεις και πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα ότι ο πατέρας σας είναι θύμα μιας βάναυσης ε, πολύ στιγνής και σκληρής μηχανής, μηχανής που συνθλίβει τους ανθρώπους. Ε, θέλουν να αλλάξουν την αυτόνομη περιοχή των Ιγούρων που είναι ιδιαίτερη. Μιλάμε για μια ειδική περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας ολόκληρης μειονότητας, μιας ολόκληρης κοινότητας. Αυτό το είδους η καταπίεση πάει πολύ πιο μακριά και ο πατέρας σας γνωρίζει την καταπίεση ως Ουιγούρος, ως πανεπιστημιακός και πνευματικός άνθρωπος και μέλος της ελίτ αυτής της κοινωνίας και ως ένας άνθρωπος θαραλέος που έχει αντισταθεί στο σύστημα. Πραγματικά λοιπόν σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε ε, και για την παρουσία σας και όσα είπατε και ευχαριστούμε και για τον πατέρα σας, ο κύριος Τέρτς. Καλησπέρα σας. Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά που ήρθατε και για τις απενεμήθεις των πατέρα σας στο βραβείο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Αφορά όλα αυτά τα θύματα του καθεστώτος. Καλά το είπε η κυρία Φοντίγα. Θύματα ολοκληρωτισμού. Τα θύματα είναι μια μειονότητα και εκεί μαζί και κάποιοι που αντιστέκονται, ο πιο εξέχων από του είναι ο πατέρας σας, που είναι στη φυλακή σε Ισόβια, με αυτή την δίκη παροδία. Και εδώ και δύο χρόνια, όπως είπατε, έχει εξαφανιστεί, κανείς δεν ξέρει την τύχη του, πρόκειται για αφόρητη κατάσταση. Τι γίνεται στην Ευρώπη πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε, είμαστε ε, ε, ανίκανοι ενώπιον αυτού του Κινέζου γίγαντα. Αλλά θα πρέπει να του αντιμετωπίσουμε και έχει διαπιστωθεί ότι να, σε κάποια θέματα ιδίω ε, πνευματική ιδιοκτησία καταφέρνουμε. Γίνονται βήματα πρόοδου και στέκεται και απαντά όταν υπάρχουν επιχειρήματα βάσιμα και όταν ε, κατησχύουν τα επιχειρήματα υποχωρεί η Κίνα. Επομένως, θα πρέπει το ίδιο να γίνει και σε θέματα τέτοιας κατάφορη παραβίασης δικαιωμάτων όπως στην περίπτωση του πατέρα σας και όσον αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας των Ιουγούρων. Άρα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε σε αυτό το μέτωπο. Να σταματήσει να έχει επιταγή λευκό η κοινοποστώσει δεκαετίες και στα εμπορικά και σε όλα τα άλλα. Με αυτόν τον κατευνασμό, την παρέτηση όλων ενώπιον τη Κίνα. Εάν δεν υπήρχε τέτοιου είδου ε, τοπάθεια, αν σταματήσει αυτό, τότε πιστεύω ότι θα πιάσει το από αυτό το βραβείο. Και κάθε είναι για τον πατέρα σα και θα, θα ξαναγεννηθούν οι ελπίδε μα Και ευχαριστούμε που ήρθατε. Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε στην κυρία Φωτίγκα. Όχι. Ο Μπαν Κρέσπο. Για την Κούβα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια πρώτα πρώτα, μπράβο σας και για τους αγώνες που έχετε δώσει, για τους Ουιγούρους και συμφωνώ ότι μακάρι να μην χρειαζόντουσαν τέτοιου είδους ε, αναγνωρίσεις να μην ήταν ε, αναγκαίες τέτοιες κινήσεις για να μην, να μην είχαμε δηλαδή πουθενά στον κόσμο παραβίαση δικαιωμάτων ούτε στην Κίνα ούτε αλλού σε άλλες πολλές χώρες και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πολλές φορές δεν κοιτάμε το περιβόλι μας οπότε είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε το ότι πολλές φορές μας διακρίνει κάποια υποκρισία όταν ασχολούμεθα με τέτοια βραβεία. Διότι ας θυμηθούμε τι έγινε το 2015. Δώσαμε σε έναν blogger από τη Σαουδική Αραβία το βραβείο. Βεβαίως και υπήρχαν ε, παραβιάσεις δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Δεν έγινε τίποτα. Και αυτό έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις. Νασέρ Ασάφη που ήταν ε, φιναλίστ για αυτό το βραβείο από το Μαρόκο. Εμείς μετά παράλληλα κάτσαμε και ψήφισαμε υπέρ συμφωνίας με το Μαρόκο. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, διπροσωπεία. Ε, έτσι αμαυρώνονται αυτά τα βραβεία και να θυμίσω και για άλλους φιναλίστ. Μόνο Καουνταλίτσια, Πάξτον, η ε, Βραζιλιάνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, η, η ακτιβίστρια. Επομένως, τα πράγματα είναι περίπλοκα. Στη Βραζιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάτσει να διαπραγματευτεί συμφωνία με τη Βραζιλία, συμφωνία εμπορική. Μιλάμε για καθεστώ που καταβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μια που είχαμε τώρα την COP25, δεν προσυπέγραψε η Βραζιλία ούτε τη συμφωνία των ε, Παρσιών για αυτή την κατεπίκουσα κατάσταση για το κλίμα που συζητούμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και πάλι πάντως να σας συγχαρώ και ελπίζω να μην ξαναδοθεί αυτό το βραβείο και να μην έχουμε ποτέ ξανά παραβιάσεις δικαιωμάτων. Thank you. Σας ευχαριστώ. Από τους μη εγγραμμένους θέλει κανείς το λόγο. Not the case. Would you like to comment once again? Μήπως θέλετε να απαντήσετε. Yeah, we'll have a second round then. Θα έχουμε δεύτερο γύρο μετά. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα ή να συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε. Δεύτερος γύρος. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Η κυρία να Μοχάμετ. Κύριε Μοχάμετ, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο. Ε, ζητώ συγγνώμη. Καλά. Θα έρθει η ώρα σου ε, ε, Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι στιγμές που ζείτε. θα ευχόμουν να μην είχαμε αυτό το βραβείο, να μην ήσασταν εδώ να ήσασταν με τον πατέρα σας και να μην χρειαζόταν. Αλλά στον κόσμο που ζούμε χρειάζεται περισσότερο από ποτέ το βραβείο Ζαχάροφ. Και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πολύ περισσότερο από ποτέ. Και μπορούμε να είμαστε η δύναμη του καλού στον κόσμο. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι παραμείνετε δυνατοί. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό το φυλάδιο, αλλά το όνομα του πατέρα σας περιλαμβάνεται εδώ μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες όπως είναι ο Νέλσον Μαντέλα, Κόφι Ανάν, ε, Λάιλα Ιούσεφ Ζάι. Παρακαλώ να μείνετε δυνατοί. Έχετε την υποστήριξή μας, όχι μόνο των βουλευτών, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο Μεζούτ Özil, Γερμανός ε, ποδοσφαιριστής που παίζει στην Arsenal τώρα, στην Premier League, ε, ξέχουσα προσωπικότητα του ποδοσφαίρου σας υποστηρίζει. Ε, και πραγματικά ε, ρίχνουμε φως στην αδικία που ζει ο λαός σας στην Κίνα. Και υποστηρίζουμε τον Φιλ Μπάνιον και τους άλλους συναδέλφους, ε, εκείνοι βέβαια πολύ περισσότερα χρόνια από μένα. Έχω να σας ρωτήσω, αν είχατε ελεύθερη πρόσβαση εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια θα ήταν τα τρία πράγματα που θα μας ζητούσατε να κάνουμε. Τα τρία πράγματα. Και ατομικά, αλλά και ως Κοινοβούλιο και ως Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Ορμπάν Κρέσπο, σας παρακαλώ σβήστε το μικρόφωνο σας, γιατί το ξεχάσατε ανοιχτό. Ευχαριστώ κύριε. Τα τρία πράγματα που θα ζητούσατε από το Κοινοβούλιο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Έχω κάποια αιτήματα, τα είχα στο μυαλό μου. Αλλά όπως είχε πει, επειδή εγώ μεγάλωσα τον μικρότερο αδερφό μου, ε, του άλλαζα τις πάνες και του τίμαζα το γάλα του, έχουμε πολύ στενούς δεσμούς, αδερφικούς δεσμούς. και είναι πολύ μικρό, αλλά πραγματικά έχει προβλήματα καρδιά με την καταστολή αυτή από την κινέζικη κυβέρνηση. Είναι 13. Σε 2,5 χρόνια θα πρέπει να πάει στο Λύκειο. Βάσει τη κινέζικη πολιτική θα έχει δυσκολίε. Δυσκολίε να πάει στο Λύκειο στην πόλη που ζει. Θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στην περιοχή των Ουγγουρών για να πάει Λύκειο. Και δεν Νομίζω ότι θα είναι ασφαλή εκεί. Κανεί από την οικογένειά μου δεν το πιστεύει. Οπότε το πρώτο που θα ήθελα να, που θα ζητούσα από το Ευρωκοινοβούλιο είναι να προσφέρει στον αδερφό μου μια ευκαιρία. Να βοηθήσει τον αδερφό μου να πάει σε οποιοδήποτε σχολείο, οποιοδήποτε λύκειο στο Πεκίνο που κατοικεί, ε, χωρίς να φοβάται. Αυτό θα ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, θα ήθελα το κοινοβούλιο να βοηθήσει εμένα την ίδια. Να μάθω ε, πού βρίσκεται ο πατέρας μου, αν είναι ασφαλής, αν μπορούσα να τον δω κιόλα σε βίντεο και να λέει την ημερομηνία της ημέρας και μια κουβέντα, μια λέξη που να λέει ότι είναι καλά. όχι το μόνο βίντεο που έχω πριν από πέντε χρόνια. Πραγματικά αυτό θα ήταν φανταστικό. Και το τρίτο, θα ήθελα το κοινοβούλιο να σκεφτεί το θέμα των κυρώσεων. Κυρώσεων για την κινέζικη κυβέρνηση και το θέμα των ε, καταβλισμών, των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτά μου έρχονται στο μυαλό. Συνάδελφοι, Άλλος ένας συνάδελφο έχει ζητήσει το λόγο, η κυρία Γενμπού. Κάποιος άλλος που δεν έχω δει. Okay, then, these two, Madame Yenbu. Merci. Η euh, ναι, κυρία Γενμπού. καλησπέρα σας κυρία Ιλάμ. Χαιρόμαστε που είστε σήμερα μαζί μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαιρετίζω το θάρρο σας και του πατέρα σας και όλων των Ιγούρων που καθημερινά αγωνίζονται. Όταν σκέφτεται κανεί την Κίνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατευθείαν σκέφτεται τη μειονότητα των Ουιγούρων αλλά και των Θιβετιανών, τον λαό του Θιβέτ. Ε, Προβληματικέ καταστάσει, διαφορετική η μία από την άλλη, αλλά ε, τελείω ιδιαίτερε. Αυτό που έχετε κοινό είναι το κεντρικό πρόβλημα που είναι η κινέζικη κυβέρνηση και η παραβίαση των δικαιωμάτων σα. Κατά την άποψή σα, υπάρχει ένα τρόπο να ε, συμπαραταχθούν οι δύο αγώνε και τι θα έπρεπε να γίνει προ αυτό το σκοπό. the last question? Θα μπορούσε η μετάφραση να, να επαναλάβει την τελευταία ερώτηση. Ναι, ε, αν θα μπορούσαν να συγκλίνουν οι δύο αγώνες. Οι Φιβετιανοί με τους Ιγούρους και το Χονγκ και την Ταϊβάν. Και εάν ναι, πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Um, I Προσωπικώς δεν έχω ποτέ έρθει σε επικοινωνία με ανθρώπους από το Χονγκ Έχω φίλους από την Ταϊβάν. Νομίζω ο κόσμος στο Χονγκ Κόνγκ, όπως και ο Ιγούρη ε, πραγματικά ε, υποφέρουν ε, με παρα... λόγω παρόμοιων προβλημάτων. Βεβαίω το Χονγκ είχε την τύχη να έχει τι τελευταίε δεκαετίε πρόσβαση σε ελεύθερα μέσα, προτού η κινέζικη κυβέρνηση τους βάλει όλους σε στρατόπεδα, πρόλαβαν να πούν τις ειδήσει που είχαν να πούν. Και πραγματικά θαυμάζω τον κόσμο που βγαίνει και διαμαρτύρεται, που κατεβαίνει και διαδηλώνει. Και Πραγματικά χαίρομαι για αυτό το θάρρος τους. Ε, εύχομαι και οι Ουιγούροι να είχαν αυτή τη ε, δυνατότητα, να βγουν στους δρόμους μαζί. Όμως, μόλις συγκεντρωθούν 10 άτομα στο ίδιο σημείο από την κυβέρνηση της Κίνας, το θεωρούν εξτρεμιστική ενέργεια. Νομίζω όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό. Δεν αγωνιζόμαστε κατά της Κίνας. Δεν έχουμε αγώνα κατά της κινέζικης κυβέρνησης. Ε, η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα, γιατί επιβάλλει σε όλους τους πληθυσμούς, χριστιανικές ομάδες, τους ίδιους τους πολίτες της χώρας, όποιος κι αν είναι, ε, τους καταστέλει. Όχι η κινέζικη κυβέρνηση, όχι η Κίνα αυτή καθεαυτή, αλλά ο τρόπος μεταχειρίζεται τους πολίτες της. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Και όπως είπα σε μια από τις προηγούμενες απαντήσεις μου, δεν είναι πολιτικό, είναι θέμα ανθρωπιστικό. Πραγματικά η κινέζικη κυβέρνηση πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Εάν όλες οι χώρες τους λένε κάνατε λάθος, δεν βοηθάει σε τίποτα να μην παραδέχονται τι έγινε και να εθελοτυφλούν και δεν μπορούν να ε, αρπάζουν την αλήθεια από τους πολίτες τους. Ευχαριστώ. Τελευταία η κυρία Χέρτσπεργκερ. Ευχαριστώ. Χέρτσπεργκερ Φοφανά. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ από όσα μας είπατε για τον πατέρα σας και από τα βάθη του κελιού του πραγματικά θα είναι περήφανος που έχει μια κόρη σαν και εσάς, που αψηφά τον κίνδυνο. Γιατί είπατε τι κινδυνεύετε να πάθετε εάν ε, έρθετε σε επαφή με τον πατέρα σας. Πράγμα σχεδόν αδιανόητο για μας αυτή τη στιγμή όπου μπορούμε να τηλεφωνήσουμε και να μιλήσουμε με όποιον θέλουμε και η οικογένειά σας τα φοβάται να έρθει σε επαφή με τον πατέρα σας. Είναι βασανιστήριο αυτό, ηθικό βασανιστήριο για σας. Η απονομή του βραβείου αυτός ε, μένει ότι υποστηρίζουμε και όλους τους άλλους αποστόλους της αλήθειας και της ε, ελευθερίας ε, όσοι θέλουν να ζήσουν με ειρήνη, να ζήσουν την πίστη τους ε, με βάση τις δικές τους πεπιθήσεις και τις θρησκευτικέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτεί φόρο τιμή στον πατέρα σας που είναι άνθρωπος του διαλόγου και το μοναδικό του έγκλημα είναι που χρησιμοποίησε το λόγο. Το λόγο, ο λόγος δεν είναι όπλο που πονάει ε, που πληγώνει, αλλά είναι ένα όπλο που θα υποχρεώσει την κινέζικη κυβέρνηση να ανακρούσει πρίμνα. Ακούσαμε τις τρεις ευχές που κάνατε. Εγώ που είμαι μια ταπεινή βουλευτής, μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υλοποιήσουμε, ε, ε, να εκπληρωθεί μία ευχή για τον αδελφό σας. Πραγματικά με συγκινεί αυτό. Κάθε χρόνο εορτάζουμε την ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Και υποθέτω ότι και στην Κίνα εορτάζουν την ημέρα του παιδιού. Και θα μπορούσαμε έτσι εμείς να βοηθήσουμε, τουλάχιστον, να μπορέσει ο αδελφός σας να ζει όπως όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ζουν τα 13 χρόνια. Να βγαίνουν στο δρόμο, να παίζουν μπάλα, ε, να κάνουν τις ανοησίες και τις βλακίες που κάνουν τα παιδιά. Και αυτό θα ήταν ίσως το μεγαλύτερο δώρο που θα, και το ωραιότερο που θα μπορούσαμε να χαρίσουμε και στον πατέρα Ευχαριστώ. I just Κυρία ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, δεν βλέπω κάποιος άλλος να θέλει το λόγο. Θέλετε μια τελευταία δήλωση. Όχι, απλώς να ευχαριστήσω όλους όσοι είστε εδώ στην αίθουσα. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και που έχετε την ε, προθυμία να μ' ακούσετε και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας και να υποστηρίξετε τον πατέρα μου. Πραγματικά το εκτιμώ ε, βαθιά. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ και την κυρία Ιλάμ. Πολύ προσωπικά, πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε και ε, χαιρετίζουμε ε, το θάρρος του πατέρα σας αλλά και το δικό σας που ήρθατε προσωπικά εδώ. Εξ ονόματος της Μαρία Γενά και του Τόμας Τομπέ ε, θα ήθελα να κηρύξω το πέρα της συνεδρίασης. Συνάδελφοι, ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12 στην Ολομέλεια για την τελετή απονομής. Ευχαριστώ και πάλι. Λήξη συνεδρίασης.